Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε παρακαλώ τις εργασίες μας. Με βάση την ημερήσια διάταξη, την οποία έχετε λάβει στις 26 Οκτωβρίου, ορίζεται ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης η έγκριση αυτής. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω αν υπάρχουν παρατηρήσεις επί της ε, ημερήσιας διάταξης. Μάθαμε ότι είναι λίγο νωρίς για να συζητήσουμε για τα αποτελέσματα της Προεδρίας του Συμβουλίου. Κανονικά έπρεπε να γίνει μια συνάντηση με τον πρόεδρο, την πρόεδρο Μάλστρουμ, αλλά σήμερα δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Επομένως, ο συνάδελφός μας, ο κύριος Νταφ, μ' ακούτε? Δεν μ' ακούτε? Funziona, Σας έλεγα λοιπόν ότι η πρόεδρος κυρία Μάλστρομ δεν θα μπορέσει να παραστεί και επομένως δεν μπορούμε να ενημερωθούμε πιο συγκεκριμένα για τις ε, εξελίξεις ε, των εργασιών του Συμβουλίου. Ο συνάδελφός μας λοιπόν ο κύριος Νταφ μου είχε ζητήσει να ξεκινήσω εγώ τη συζήτηση για αυτό το θέμα. Φυσικά είμαι στη διάθεσή σας να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό που ξέρουμε στην πραγματικότητα είναι μόνο η επίσημη ανακοίνωση στον τύπο από πλευρά του Συμβουλίου. Εκεί εκφράζεται η πεποίθηση του Συμβουλίου ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα θα εγκριθεί μέχρι το τέλο του 2009 και εκφράζει την ικανοποίησή του. Μάλιστα, σήμερα το πρωί μάθαμε ότι το τσεχικό συνταγματικό ε, δικαστήριο απέρριψε τα όποια τους λόγους αντισυνταγματικότητας της συνθήκης της Λισαβόνας και επομένως περιμένουμε την υπογραφή από τον Τζέχο Πρόεδρο σε λίγες μέρες. Ίσως ε, στην αρχή μάλιστα της επόμενης εβδομάδας. Όλα τα στοιχεία κατατείνουν προς αυτό. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο να πει κάτι. Ο κύριος Μέντες Τεβίγκο. Εγώ εκ μέρους ομάδας μου θα ήθελα να εκφράσω την απέραντη ικανοποίηση που αισθανθήκαμε και για τα απορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και για την λύση που δόθηκε από το Ζεχικό Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της προσφυγής του Προέδρου, που ήταν ούτως ή άλλως αλλοπρόσαλη. Αλλά αυτή είναι η Ευρώπη. Αναζήτηση συμβεσμών, συμβαστικών λύσεων προκειμένου να ανεβρεθεί συμφωνία. Αυτή είναι πολύ χαρμόσυνη είδηση, την αναμέναμε όλοι, αλλά επιτέλους επιβεβαιώθηκε και για τρίτη φορά το Τσεχικό Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόπειρα κήρυξη συνταγματικότητα της συνθήκης. Εμεί είμαστε υπέρ και τη συνταγματική συνθήκη και τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γι' αυτό και για όλου εμά ε, σήμερα είναι μια πολύ ευτυχή ημέρα. Και αυτό παρακαλώ να σημειωθεί στα πρακτικά, γιατί φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία των ε, πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, πιστεύει, ακόμη και αν είναι κατά των της ίδιας συνθήκης Λισαβόνας, ε, πιστεύει ότι το έργο που επιτέλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 2000 μέχρι σήμερα τελικά απέδωσε καρπούς. Και αυτό που είναι να αφισβείται, είτε μας αρέσει η συνθήκη είτε όχι, είναι ότι το Κοινοβούλιο είναι ένα από τους βασικούς θριαβευτές αυτής της συνθήκης της Λισαβόνας και ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών μπορούμε να αισθανόμαστε ικανοποίηση γιατί στο μέλλον θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Πολύ κερια αυτές οι παρατηρήσεις. Ο κύριος Γιαρέγκουι. Sí, και εγώ, εκ μέρους ε, των σοσιαλιστών, θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη ικανοποίηση που μας προκάλεσε η σημερινή αυτή είδηση. Όχι μόνο όμως για το δικαστήριο, γιατί και το Συμβούλιο το περασμένο Σαββατοκυριακό υιοθέτησε μια πολύ σημαντική απόφαση, γιατί επέλυσε ένα πολύ περίπλοκο πολιτικό ζήτημα με την απόφασή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αισθανόμαστε λοιπόν ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί επιτέλους ε, ε, θα κυρωθεί η συνθήκη κατά πάσα πιθανότητα το Νοέμβριο και θα τεθεί σε ισχύ από τον επόμενο μήνα. Και η έχουμε και την πολιτική απόφαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που τις επόμενες μέρες θα διαλέξουν τον πρόεδρο του Συμβουλίου και τον είπα εκπρόσωπο και ο πρόεδρος της Επιτροπής ο κύριος Μπαρόζο θα σχηματίσει τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμεί σήμερα θα εγκρίνουμε το νέο κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οριστικά πια θα τεθεί σε ισχύ από την 1η του 2010 και θα σημάνει την ε, απαρχή μιας ε, νέας πορείας και μιας νέας όθησης ε, στο παλιό όνειρο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και της εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε αυτό συνδυάζεται με μια εμφανή πολιτική ανάγκη, γιατί αν πριν από 60 χρόνια το ευρωπαϊκό όραμα και όνειρο γεννήθηκε ε, με την επιθυμία να αποκατασταθεί η ειρήνη πάνω στα ερήπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα η ευρωπαϊκή συζήτηση είναι συζήτηση να ζει κανεί ή να μη ζει, σαν το δίλημα του Άμλετ στην Ευρώπη. Υπάρχει η επιθυμία να ακούγεται ενωμένη η φωνή της σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, να έχει δικό βάρος στο νέο γεωστρατηγικό και οικονομικό παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα, ακούει, θα ακούγεται τη φωνή της, θα είναι ενωμένη και όχι διχασμένη, γιατί χωρίς ενωμένη Ευρώπη δεν υπάρχει καν Ευρώπη. Αυτή είναι η συζήτηση των τελευταίων ημερών. Και οι τελευταίες εξελίξεις και οι σημερινές και τις προηγούμενες εβδομάδες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να ξεκινήσουμε αυτή τη νέα πορεία που πολύ σωστά είπε ο κύριος Μέντες Δεβίκο, ξεκίνησε πριν από μία δεκαετία περίπου αλλά πέρασε από 40 κύματα. Γιατί μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν ήμασταν βέβαιοι ότι θα καταφέρναμε να ξεπεράσουμε τα κολλήματα και τις κοπέλους που καθημερινά έβρισκαν μερικοί σε αυτό το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν αισθανόμαστε αυτή την απέραντη ικανοποίηση για τι τελευταίε εξελίξει. Αλλά αισθανόμαστε και κάποια απογοήτευση γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Σαββατοκύριακου επισήμανε εύγλωτα τα σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω των κλιματικών αλλαγών. Και παρόλο που στα πορίσματα το Συμβούλιο, το Συμβούλιο ε, αναγνώρισε αυτά τα προβλήματα, έλαβε μία θέση έναντι του της διάσκεψης κορυφής Κοπεχάγης που μάλλον είναι ανέφικτη να υλοποιηθεί. Πάντως ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μα δημιούργησε δυστυχώ την ανησυχία ότι κατά πάσα πιθανότητα η διάσκεψη κορυφή Κοπεχάγη δεν θα σημάνει πρόοδο ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και παρά τις εσωτερικές δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και την ε, υπόσχεση βοήθειας των αναπτυσσομένων χωρών να ενστενιστούν το Κιώτο και να περιορίσουν τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα, πολύ φοβάμαι ότι παρόλα αυτά σημαντική πρόοδος στην Κοπεχάγη δεν θα σημειωθεί για το κλίμα. Και αυτή είναι η ανησυχία που προέκυψε από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε την ε, περίπλοκη μακροοικονομική συζήτηση που γίνεται αυτή τη φορά στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ανάκαμψης και τη Ευρωπαϊκή οικονομία και τη παγκόσμια κατάστασης, αλλά έχουμε και δύο πολύ σοβαρά προβλήματα στη μακροοικονομική μας πραγματικότητα. Έχουμε μία καλπάζουσα ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο έλαβε χώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έδωσε μια είδηση με την επίλυση του σοβαρού πολιτικού προβλήματος και μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία ε, και μια τρίτη χώρα αποσπάστηκε από το χάρτη των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά παρόλα αυτά το Συμβούλιο έδωσε μια λύση σε ένα κεφαλαιόδες πρόβλημα αλλά δημιούργησε και κάποιες ανησυχίες για αυτά που σας είπα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και την αδυναμία ως προς, την, ως το, προς το περιορισμό της ανεργίας. Ο κύριος Νταφ θα μιλήσει τώρα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σταθώ στη συνταγματική πλευρά της συζήτησης που προέκυψε από τη συνάντηση του Συμβουλίου. Δεν έχουμε μόνο τα συμπεράσματα της Προεδρίας, αλλά και το σχέδιο πρωτοκόλλου, το οποίο θα προσαρτηθεί στο πρωτόκολλο υπαριθμών 30 για τη Τσεχία. Με έκπληξη είδα ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί πίστευα ότι ο πρόεδρος Κλάους από πειράτο να πετύχει ένα πρωτόκολλο το οποίο θα καθορίσει τις ρήτες ιδιοκτησίας στη χάρτα και όχι τις ρήτρες για τα κοινωνικά θέματα που υπάρχουν στη χάρτα. Θα ήθελα να είχα την ευκαιρία να θέσω κάποιες ερωτήσεις στην Προεδρία για τη σημασία που θα πρέπει να δώσουμε σε αυτό το προσχέδιο, σε αυτό το προτινόμενο σχέδιο πρωτοκόλλου. Δεύτερον, παρότι και εγώ είμαι ικανοποιημένος για την απόφαση του δικαστηρίου στον Πρνό, Ακόμα δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι εγγυήσει ότι ο πρόεδρος Κλάς θα υπογράψει το κείμενο. Δεν υπάρχει τίποτα γραπτό και τίποτα σχετικό στα συμπέρασματα της Προεδρίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να μην εκφράσουμε τώρα την ικανοποίησή μας για το θέμα της συνθήκης. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να έχουμε όλα τα εχέγγυα, μέχρι να έχουμε την υπογραφή του κ. Κλάς. Ωραία. Μετά τον κύριο Νταφ, ο κύριος Ζάιερ. Thank you very much, uh, President. We are just a uh, ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, λίγα λεπτά μόλις ε, απέχουμε από την υπογραφή της Συνθήκης Λισαβόνας, οπότε θα τεθεί ενισχύ και θεωρώ πως άλλο ένα τεχνητό εμπόδιο παραμερίστηκε στην διαδικασία, αλλά συμφωνώ με τον τελευταίο μιλητή, τον κύριο Νταφ, πως ε, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν έχουμε εγγύησει για την τελευταία πράξη, την υπογραφή δηλαδή του Τσέχου Προέδρου. Πράγματι εδώ είναι το σωστό μέρος να το συζητήσουμε γιατί εδώ όπως ξέρετε έγινε και η συντακτική συνέλευση και πολλοί συνάδελφοι θα ήθελα να πούν πόσο σημαντική είναι η συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ όμως θα ήθελα να θίξω κάτι άλλο που ανέφερε ήδη ο κύριος Νταφ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέλαβε μία δέσμευση για το opt-out της τσεχικής δημοκρατίας από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το κοινοβούλιο μας έχει κάποια, υιοθετήσει κάποια ψηφίσματα στα οποία εκφράζουμε την λύπη μας για το ότι δύο άλλες χώρες επίσης δεν ε, υπέγραψαν τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων γιατί εμείς σταθερά είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σχετικής χάρτας. Έχουμε λοιπόν σταθερή θέση. Οπότε δεν είμαι ικανοποιημένο για το ότι εξαιρείται η τσεχική δημοκρατία και ακόμη λιγότερο για το ότι αυτό γίνεται με το πρόσχημα που ανέφερε ο πρόεδρος ο κύριος Κλάους και τα επιχειρήματα που είπε ότι δηλαδή φοβάται πως ε, τα διατάγματα μπένες ε, ε, εξακολουθούν να έχουν κάποια αποτελέσματα για κάποια ισχύ. Να σας θυμίσω πως τα διατάγματα μπαίνες, τα 13 αυτά, βασίζονται σε συλλογική ευθύνη, σε διακριτική μεταχείριση, σε εθνοτικό μίσος. Οπότε δεν είναι αποδεκτό αυτό το επιχείρημα. Π.χ. ούτε στη χώρα μου αλλά και στη Γερμανία, την Αυστρία και αλλού. Δεν είναι αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα το οποίο αναφέραμε και πρέπει να το τονίσουμε. είπα αυτή την έννοια, εάν ήμουν βουλευτής στο Εθνικό Κοινοβούλιο, δεν θα υπερψήφιζα την εξαίρεση της Τσεχίας, ειδικά με βάση αυτά τα επιχειρήματα, γιατί αυτό είναι απαράδεκτο. Γνωρίζω π.χ. την θέση του εθνικού μου κόμματος ε, στην Ουγγαρία πως δεν πρόκειται να υποστηρίξουν κάποια αλλαγή της συνθήκης ε, που θα συμπεριλαμβάνει αυτή την εξαίρεση της Τσεχίας με το πρόσχημα ότι θέλουν να προστατευτούν ε, από τις νομικές συνέπειες των διαταγμάτων Μπένες. Οπότε πρέπει να το γνωρίζουμε και βεβαίω να πούμε ω Κοινοβούλιο πω είμαστε ικανοποιημένοι για τη συνθήκη τη Λισαβόνα, αλλά ταυτόχρονα είμαστε υπέρ τη χάρτα αυτή και να εφαρμοστεί σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γιατί πήρα το λόγο. Ο συνάδελφο είπε ότι πρέπει να καταγράψουμε στα πρακτικά ότι η σημερινή μέρα είναι μια ευτυχισμένη μέρα και το θετικό είναι ότι η συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί οπωσδήποτε σε ισχύ. Αλλά δεν είναι δεδομένο ότι συμμεριζόμαστε όλοι αυτή την, αυτό το αίσθημα και αυτή την ιδέα. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το κοινοβούλιο, όπως λέγεται εδώ, ότι εκπροσωπεί ολόκληρο τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Σκεφτείτε τις προσφυγές που έχουμε ε, στα συνταγματικά δικαστήρια στη Γερμανία Φερρυπίν. Αυτές ε, οι προσφυγές ε, σε ένα ανώτατο ε, όργανο όπως το συνταγματικό δικαστήριο δείχνουν ότι η όλη διαδικασία είναι αμφιζητήσιμη όχι μόνο για την συνθήκη της Λισαβόνας. Εκεί καταλαβαίνω τα επιχειρήματα υπέρ της συνθήκης. Αλλά η διαδικασία δεν νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που μας εξασφαλίζει τη δημοκρατία. Ε, αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι να ακούσουμε τη φωνή του Βρετανικού λαού. Και θέλουμε να ε, υιοθετηθεί άρον-άρον αυτό το, αυτή η συνθήκη, ούτως ώστε να μην μπορέσουν να κάνουμε το δημοψήφισμά του στη Βρετανία. Γι' αυτό ακριβώς Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι σοβαρή αυτή η διαδικασία. Και θα ήθελα αυτό να καταγραφεί στα πρακτικά. Όχι ότι είναι αυτή η αίσθηση και η άποψη της πλειοψηφία των βουλευτών, αλλά ότι είναι η δική μου άποψη αυτή. Και επίσης, αυτό το opt-out, αυτή η παρέκκληση σε σχέση με τη χάρτα, ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τη νομική υπηρεσία να διερευνήσει σε ποιο βαθμό πρόκειται για μια εξήγηση για μια διευκρίνηση, για ένα πρωτόκολλο. Τι ακριβώς υποσχεθήκαμε στην Τσεχία και στον Βάκλαβ Κλάους. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω ε, να το ξέρουμε αυτό για να δουλέψουμε σε στέρεες νομικές βάσεις. Και αυτό βεβαίω ε, στο βαθμό ε, που θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, θα επικυρωθεί δηλαδή η συνθήκη και τελικά θα τεθεί σε ισχύ. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε εκ των προτέρων. Η κυρία Γκουρμάη. Βεβαίως ε, χαιρόμαστε για την απόφαση του τσεχικού συνταγματικού δικαστηρίου, αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που έδωσαν το, το πράσινο φως. Βεβαίως ε, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί πρέπει να είναι σαφές πως ε, ο κύριος Κλάους ξεκαθάρισε πως θα υπογράψει. Και δεν νομίζω τώρα πως μπορεί να ζητήσει τίποτα άλλο από τις υπόλοιπες 26 ε, χώρες που έχουν ήδη υπογράψει και ακόμα αναμένουμε το τι θα γίνει όσον αφορά και την επόμενη Κομισιόν γιατί θέλουμε να ακούσουμε και τους υποψήφιους και βεβαίως είναι σαφές Όπως είπε και ο συνάδελφος από την Ουγγαρία όσον αφορά την χάρτα, δύο κράτη-μέλη είχαν την ευκαιρία να μην την αποδεχτούν. Είχαν την δυνατότητα δηλαδή να εξαιρεθεί και να εξαιρεθεί και η Τσεχία πολύ νωρίτερα. Οπότε ας είμαστε λογικοί. Νομίζω πάνε καλά τα πράγματα για την συνθήκη της Λισαβόνας και ελπίζω ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ε, προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε αλλά πρέπει να σεβαστούμε βεβαίω και τα 15 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών και συμφωνώ εδώ πέρα με τον συντονιστή του ΕΛΚΑ Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ σκληρά, πρέπει λοιπόν τώρα να γίνει πραγματικότητα. αλλά παρόλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πέρασε πολύ καιρός για να τα καταφέρουμε εδώ πέρα, είτε το πούμε συνταγματική συνθήκη είτε Λισαβόνα. Σχεδόν μια δεκαετία. Και αυτό μας λέει κάποια πράγματα, έτσι, αν το δούμε μακροπρόθεσμα με μια ιστορική σκοπιά. Εγώ έχω την αίσθηση πως αυξάνεται η διακυβερνητική προσέγγιση, ενισχύεται, πως ε, η αντίθεση στην ευρωπαϊκή ενοποίηση αυξάνεται και θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ρεαλιστικά η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση λύνει πράγματα που δεν μπορούν να λυθούν με την διακυβερνητική προσέγγιση. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που μπορούν να λυθούν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως έτσι και πάλι μακροπρόθεσμα ιστορικά αν το δούμε πρέπει να δούμε πως δεν έχουμε πια τα προβλήματα εκείνα στην Ευρώπη τα οποία καταδυνάστευαν τις ε, διεθνείς σχέσεις ε, στο Μεσοπόλεμο και οδήγησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε από αυτή την ε, άποψη είναι μια μεγάλη επιτυχία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε εάν το δούμε έτσι όσο περισσότερες εξαιρέσεις έχουμε τόσο χειρότερα είναι τα πράγματα. Και ειδικά μια εξαίρεση με βάση την αρχή της συλλογική ενοχής είναι η πιο απαράδεκτη από όλες. Grazie. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πρέπει να πω και εγώ δύο λόγια, εν κατακλείδη, ε, για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Εγώ εμπιστεύομαι ότι θα τελεσφορήσει όλη η διαδικασία της ε, κύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας. Μου φαίνεται πραγματικά παράλογο το να μην ε, ολοκληρωθεί επιτυχώς. Δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό ότι θα αναβαγίσει όλη η διαδικασία εξαιτία του Προέδρου της Τσεχίας. Προκύπτουν λοιπόν αισθήματα ικανοποίησης αλλά και κάποιες ανησυχίες ε, γιατί καταγράφτηκαν όλες οι δυσκολίες της ε, διαδικασίας και εκφράστηκαν τους συναδέλφους. Εγώ, κοιτάξτε, έχω διαβάσει πολλές φορές τη συνθήκη της Λισαβόνας και 7 φορές μάλιστα. Ε, αναφέρεται στη συνθήκη η λέξη φάση. φάση. Η συνθήκη της Λισαβόνας επίσης πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι μια τελική στιγμή. Είναι μια φάση. Αυτή καθε αυτή η Λισαβόνα είναι μια φάση. Επομένως πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν είναι τέλεια η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει να το ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε αυτό το βήμα. Ακόμα και οι παρεκκλήσεις της Πολωνίας, της Ιρλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τσεχίας τώρα, τελευταία. Δεν, θα, δεν μπορώ να αρνηθώ ότι συνιστούν ε, κάποιο κίνδυνο. Αλλά από την άλλη ε, δεν συνιστούν ε, κανόνες, αλλά κάποιες διασαφήσεις. Κάποιες διασαφήσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι τόσο ανησυχητικές. Σε ό,τι αφορά τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεωρεί ως σημείο αναφοράς. Και επιπλέον όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κύρωσαν ως κράτη τη σύμβαση του ΟΗΕ για την διαφύλαξη των θεμελιδών δικαιωμάτων. Τώρα, για την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα ήθελα να υπάρξει κάτι έτσι το τυπικό, ε, που θα είναι και οριστικό. Νομίζω ότι υπάρχουν λόγοι αισιοδοξία. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να χαιρετήσω κάποιους διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχίας ε, που είναι παρόντες σε αυτήν την αίθουσα. Τους χαιρετίζω, του εύχομαι να τα καταφέρουν, να υλοποιήσουν τις ελπίδες τους και να συνεισφέρουν έτσι θερμά και έντονα ε, στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ας περάσουμε τώρα στις υπόλοιπες ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Για αυτές τις ανακοινώσει του Προέδρου θα περιμένω τη συνεδρίαση των εκπροσώπων των διαφόρων ομάδων που θα κάνουμε μετά το πέρας της δική μα συνεδρίασης. Έχουμε διάφορα σημεία στη μέση διάταξη για του συντονιστέ λοιπόν των διαφόρων πολιτικών ομάδων και αύριο το πρωί όταν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής θα σα πω ότι προέκυψε από τη συνεδρία των συντονιστών. Επομένω, τώρα θα μπορούσαμε να περάσουμε στο τρίτο σημείο τη ημερησία διάταξη, που είναι η προσαρμογή του κανονισμού στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Εμεί ήδη συζητήσαμε τι τροπολογίε που παρουσιάστηκαν στο σχέδιο έκθεση του κυρίου Μάρτιν. Έχουμε μπροστά μας και τις τροπολογίες της έκθεσης που είχε εγκριθεί τότε, καθώς και τις νέες τροπολογίες του κυρίου Μάρτιν. Ξέρω όμως ότι έγιναν και επαφέ για να παρουσιαστούν και συμβαστικέ τροπολογίες. Και τελικά ξέρω ότι θα υπάρξουν και προφορικές τροπολογίες. Νομίζω λοιπόν ότι όταν φτάσουμε στην ψηφοφορία των συμβαστικών τροπολογιών και των προφορικών τροπολογιών, καλό θα ήταν οι συντάκτε να μας, εξηγήσουν ακριβώ περί πρόκειται. Νομίζω ότι πολλές από αυτές τις τροπολογίες Μπορούμε να τι ψηφίσουμε συλλήβδιν. Και καθώ θα ψηφίζουμε θα κάνω και συγκεκριμένη πρόταση. Δεν ξέρω αν πριν περάσουμε στην εμφορία οι υπεύθυνοι των ομάδων θα ήθελαν να κάνουν κάποιε δηλώσει για να διευκρινίσουν τι θέσει του, ή όχι. Παρακαλώ, ο κύριο Κόξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία 60 του κυρίου Μπροκ, την οποία απέσυρε. Πρέπει να πω. Θα εξέφραζα την απογοήτευσή μου για το ότι απεσύρθη. Γιατί αυτό θα σήμαινε πως οι κανόνες που αφορούν το καθεστώς των μελών θα συζητούνταν στο κοινοβούλιο, δηλαδή δημόσια. Και είναι λυπηρό να αποσύρεται μια τροπολογία που ενισχύει τη διαφάνεια. Χωρίς εξήγησε. Ελπίζω λοιπόν να επανέλθει στην τροπολογία και θα ήθελα να ενθαρρύνω τον κύριο Μπρόκ να την επανυποβάλει. Εδώ στην πρώτη, πρώτη. Ο κύριος Μάρτιν, ο εισηγητής, έχει το λόγο. Θα είμαι λακωνικότατος, κύριε Πρόεδρε, για να μην καθυστερήσουμε στην έναρξη ψηφοφορίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ρίσαρ Κόρπετ πάντως για την προεργασία που ήταν πραγματικά τεράστια. Κανονικά, έκθεση Κόρπετ θα πρέπει να λέγεται. Και η αρρωγή που μου παρήχε τον τελευταίο καιρό ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και για τεχνικά και άλλα θέματα. Ευχαριστώ και τις πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία τους που πραγματικά ήταν αγαστή καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κύριου Κόξ, αφορούν ένα ουσιαστικό θέμα της Λισαβόνας. Δεν θέλω να προδικάζω τα όσα θα πει ο κύριος Μπροκ, αλλά σε ό,τι αφορά τους κανόνες του Προεδρείου, διαφώνησα με την τροπολογία επειδή αυτή δεν απορρέει άμεσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό θεώρησα ότι θα πρέπει να τύχει διαφορετικής μεταχείρισης. Και αν υπήρχαν κάποιοι τομείς ε, όπου υπήρχαν διαστάσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αλλά δεν αφορούσαν θέματα της Λισαβόνας, ε, δεν θα λαμβάνονταν υπόψη, για να γιατί δεν καλύπτονται από τη συμβαστική πρόταση. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να παρα, α, παρέμβουν, υπάρχουν. Ο κύριος Μπρόκ. Ε, Κύριε Πρόεδρε, με για την απόσυρση των τροπολογιών 60 και 61. Εγώ δεν τις έχω αποσύρει. Ίσως να υπάρχει κάποιος σωσίας μου εδώ πέρα που τις απέσυρε. Δεν ξέρω. Ίσως η Σύνοδος των Προέδρων ε, μπορεί να αποσύρει τροπολογίες χωρίς τη συμμετοχή των διαφερομένων βουλευτών. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω να ψηφιστούν οι τροπολογίες. Μάλιστα. Προφανώς κάτι δεν είχα καταλάβει καλά. Μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε και αυτές τις τροπολογίες. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Ωραία. Πολύ ωραία. Θέτω στην ψηφοφορία την τροπολογία 1, άρθρο 7, παράγραφος 2 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Άρθρο 8. Τροπολογία 60. Μπρόκ. Ποιος είναι υπέρ. Σηκώνει το χέρι παρακαλώ. Όποιος είναι υπέρ. 13 υπέρ, κατά. Οκτώ κατά, αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Ψηφίσουμε τώρα την τροπολογία 2, άρθρο 11, παράγραφος 3α. Του εισηγητή υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή και εγκρίνεται. Τροπολογία που δεν έχει αποσυρθεί και θα ψηφιστεί του Μπρόκα ε, μόνο 61 για το άρθρο 23, παράγραφος 2 και παράγραφος 2α. Υπέρ. Κατά. Έντεκα, εννιά, άποχες. Δύο εποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 62, άρθρο 23, παράγραφος 11α. Μάρτιν, Σάιερ και Νταφ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τρεις αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 3, άρθρο 36 του εισηγητή. Υπέρ παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια. κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Του εισηγητή για το άρθρο 38. Είναι συμβαστική τροπολογία. Θα ήθελα κάποιο να μα την παρουσιάσει, επειδή είναι πιο σημαντικέ οι συμβαστικέ τροπολογίε, όπω είπαμε. Α, διάβασα λάθο στον καταλογό μου. Για το άρθρο 4 μπορούμε να ψηφίσουμε, για την τροπολογία εννοεί ο πρόεδρο 4, μπορούμε να ψηφίσουμε χωρί να μα την παρουσιάσει κανεί υπέρ, κατά, αποχέ. ομόφωνα αν κρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία. Προφορική έχω γράψει εγώ ή συμβαστική τροπολογία, όπως γράφει ο καταλογός σας. Θα ήθελα οι συντάκτες να την παρουσιάσουν αυτή την τροπολογία, παρακαλώ τη συμβαστική τροπολογία 1. Μάρτιν. Ευχαριστώ. Είναι πολύ αυτή γιατί είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά χρειάζεται κάποια εξήγηση. Πρώτα απ' όλα εδώ πέρα εισάγεται... Το έχετε... Έχει μοιραστεί νομίζω στα συναδέλφους. Οπότε είχα την ευκαιρία να το διαβάσετε. Υπάρχει εδώ πέρα ένα νέο σημείο 4 που λέει Πλην των περιπτώσεων εκτάκτων ανάγκη που αναφέρονται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλου του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή δεν θα περάσει την τελική ψηφοφορία πριν την εκπνοή της προθεσμίας των 8 εβδομάδων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του πρωτοκόλου, εφαρμόζοντας ε, τις αρχές αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Εάν ε, περάσει αυτό πρέπει να έχουμε κάποιες διαγραφές. Δηλαδή το τωρινό 3, εάν το Εθνικό Κοινοβούλιο κτλ. κτλ πρέπει να διαγραφεί. Μετά. Στο σημείο 6, στη δεύτερη παράγραφο, εκεί που λέει ή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο οποιαδήποτε άλλη σύσταση που θα περιέχει προτάσεις ε, για αλλαγές σε σχέση με την αρχή της επικουρικότητας και αυτή η φράση πρέπει να διαγραφεί και στο τέλος ε, της συμβαστικής πρότασης εκεί πέρα που λέει λαμβάνοντα υπόψη οποιασδήποτε στάσεις που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Όλα αυτά θα πρέπει να διαγραφούν εάν αποδεχτούμε το 4. Κάτι άλλο που δεν έχουμε συζητήσει με τις ομάδες, αλλά συνιστός αλλαγή. Μίλησα με την νομική υπηρεσία πριν τη συνεδρίαση και μου είπαν πως εάν, ε, ο, εάν και ο κανόνας αυτός αφορά το πρωτόκολλο, ε, το σχετικό για την ε, επικουρικότητα και την αναλογικότητα κατά βάση αφορά την επικουρικότητα εξού και η λέξη αναλογικότητα γι' αυτό προτείνουμε ο τίτλος, γι' αυτό λένε πως ο τίτλος είναι λίγο παραπλανητικός και προτείνουν να φύγει η λέξη και αναλογι... και αναλογικότητα και να μείνει μόνο η λέξη επικουρικότητα. Είναι λίγο περίπλοκα, αλλά είναι νομίζω η μόνη περίπλοκη τροπολογία. Να ευχαριστώ κύριο Ντάφ. Από το έγγραφο που έχει διανεμηθεί βλέπετε ότι υπάρχουν μία-δύο προτάσεις που είναι γραμμένες ε, λιγότερο έντονα. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν διαγραφεί αυτές οι προτάσεις που φαίνονται πιο αχνά στο έγγραφο που μόλις μας μοιράσατε. Γιατί δεν προκύπτει με σαφήνεια. Α, εντάξει. Είναι κάπως μπερδεμένο, αλλά σας καταλαβαίνω. Ο κύριος Μάρτιν μπορεί να μας τα εξηγήσει καλύτερα γιατί επειδή δεν μιλούσατε στο μικρόφωνο, δεν μας μετέφρασαν διερμηνείς. Μπορείτε να επαναλάβετε την εξήγηση που δώσατε στον κύριο στο μικρόφωνο αυτή τη φορά. Ναι, συγγνώμη. Κοιτάξτε, εγώ το είχα υπογραμμίσει με τον Μαρκαδόρο, αλλά δεν βγαίνει βεβαίω στη φωτοτυπία. Είναι μία από τις ε, διαγραφές που θα προκύψουν από την αποδοχή του 4. Ζητώ συγγνώμη από του συναδέλφου για όλα αυτά, αλλά διαπραγματευόμασταν κυριολεκτικά μέχρι το παραπέντε. Τι, κολέγα Φόξ. Ναι, ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να μας εξηγήσει γιατί έφυγε από τον συμβιβασμό η πρόταση στην παράγραφο 5 της αρχικής τροπολογίας 64 ότι μια σύσταση μπορεί να κατατεθεί επίσης και από το 1 δέκατο των βουλευτών. Γιατί νομίζω πως ε, με αυτή τη συμβαστική λύση αφαιρούνται εξουσίες από το Κοινοβούλιο για να παραπεμφθούν ε, ζητήματα επικουρικότητας. Και αφαιρείται αυτό το δικαίωμα και από την Επιτροπή των Περιφερειών. Εδώ πέρα λοιπόν φαίνεται πως ε, αφαιρούνται εξουσίες να ξεκινήσει μια συζήτηση με βάση την αρχή της επικουρικότητας και θα ήθελα να ακούσω γιατί έγινε αυτό. Ναι, η Επιτροπή των Περιφερειών είναι κάτι που θα δούμε αργότερα παρακάτω στην έκθεση. Για το 10% των βουλευτών, ναι, είναι ο συμβασμό στον οποίο καταλήξαμε. Τώρα, εάν μου επιτραπεί να μιλήσω προσωπικά, ναι, εγώ ήμουν υπέρ, αλλά είναι κάτι που θα αποφασίσει η Επιτροπή. Ήταν ένα συμβασμό με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Θέλει κανεί άλλο το λόγο. Ψηφίζουμε λοιπόν την συμβαστική τροπολογία που ακούσατε. Όποιο την υπέρ να το χέρι παρακαλώ. Κατά. Πέντε. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 64 που καλύπτεται από αυτόν τον συμβιβασμό, αλλά παρόλα αυτά θα την ψηφίσουμε την τροπολογία. Την ψηφίσουμε? Όχι, καλύπτεται. Δεν χρειάζεται λοιπόν. Πάμε τότε στην ε, επόμενη τροπολογία. Η τροπολογία 64 ε, και 5 καταπίπτουν και πάμε στην τροπολογία 6 του εισηγητή, άρθρο 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 2. Εγκρίνεται. Και τώρα φτάσαμε στο άρθρο 56, παράγραφος 3. Υπάρχει μια άλλη συμβαστική τροπολογία. Καλό θα ήταν να μας την παρουσιάσετε, ο εισηγητής. Αυτή είναι απλή. Απλώς θα αναπέμπεται η μια έκθεση στην Επιτροπή μπορεί να ακολουθήσει κανονικές διαδικασίες είτε να την επαναλάβει, να την ξαναυποβάλει, είτε να μην υποβάλει καθόλου, είτε να υποβάλει μια έκθεση με τροπολογίες. Αναφέρεται στις στη διακριτική ευχαίρεια μια επιτροπή να δράσει σε περίπτωση που αναπέμπεται από την Ολομέλεια μια έκθεση πίσω σε μια επιτροπή. Ψηφίσουμε τότε την τροπολογία συμβιβασμού υπαριθμών 2. Υπέρ, κάποιος ένας υπέρασικο στο χέρι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Αυτή καταπίπτει. Έτσι. Πολύ ωραία. Τώρα θα κάνω την εξή πρόταση. Από την τροπολογία 7 μέχρι την τροπολογία 15, όχι, μέχρι και την 14 καλύτερα, μια στιγμή γιατί τα έχω μπέρδεψει εδώ πέρα, μέχρι και την 14, θα έλεγα να τις ψηφίσουμε μαζί, αν συμφωνείτε. Πρόκειται για τεχνικές προσαρμογές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, 65, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14. Ποιος είναι υπέρ, να σηκώσει το χέρι παρακαλώ, για αυτές τις τροπολογίες. Παρακαλώ. Διαγράφουμε εδώ πέρα το 9, 11 και το 13. Ναι, ναι, εντάξει, με συγχωρείτε. Ε, όποιος είναι υπέρα στο χέρι. Κατά. Αποχές. Τρεις αποχές. Εγκρίνονται όλες αυτές τις τροπολογίες. Και πάμε στην τροπολογία 66, Σάιερ. Κεφάλαιο 6α. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Όχι, αυτή καταπίπτει. Πρόεδρε, λέει ο κ. Νταφ. Νομίζω ότι επειδή μοιάζουν πολύ αυτές τις τροπολογίες και επειδή μάλλον και οι ψήφοι των υπέρ και των κατά είναι πολύ κοντά, θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι υπέρ και πώς είναι κατά. Στην προηγούμενη ψηφοφορία ψήφισαν 11 υπέρ και 10 αποχές. Μπορεί να επαναλάβουμε ψηφοφορία αν θέλετε. Όχι, λέει ο κύριος Νταφ. Δεν χρειάζεται. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Όχι, νομίζω ότι ψηφίσαμε. Εντάξει. Αν θέλει κάποιο ηλεκτρονική ψηφοφορία, α μου το πει. Να μου το ζητήσει, είναι απλό. Λοιπόν, η τροπολογία 15. Καταπίπτει, είπαμε αυτή. Και περνάμε στην τροπολογία 16, επί της οποίας υπάρχει μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Τροπολογία 16. Αφορά επίσης αυτή η προφορική τροπολογία και το, την 53. Ε, αφορά τη λέξη convention, σύμβαση. Ε, μια τεχνική προσαρμογή. Πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Γράψατε στον κατάλογό σας ότι με την προχωρική τροπολογία διαγράφουμε από το 132, το άρθρο 132 του καονισμού τη λέξη convention, τη λέξη σύμβαση. Το ίδιο προβλέπεται και για το 53, 54, συγγνώμη. Μπορούμε να ψηφίσουμε μαζί αυτές τις δύο τροπολογίες. Υπέρ, παρακαλώ υπέρ. Ο κύριος Νταφ. Με συγχωρείτε. Κι εγώ απορώ εδώ πέρα λέει πως πρέπει να διαγραφεί η λέξη. Αλλά στην ε, τροπολογία την ε, τη συμπεριλαμβάνει κανονικά. Στην τροπολογία 16 όταν περιγράφει την ε, διαδικασία σύγκλησης διακυβερνητικής διάσκεψης. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι την ε, αναγκαιότητα ε, διαγραφής της λέξης εδώ πέρα. Um, Συγγνώμη, ε, υπάρχει μια σύγχυση εδώ. Έχει κάποιο δίκιο ο Άντριου Ντάφα, αλλά δεν το εξήγησα εγώ σωστά. Νόμιζα ότι το είχαμε καταλάβει. Θα, θα διαγραφεί στο άρθρο 132. Και πρέπει να φύγει από το 132 γιατί το, το θέμα αυτό το βλέπουμε τώρα σε αυτό το νέο άρθρο του, του κανονισμού. Ε, εγώ φταίω δεν το, δεν το εξήγησα σωστά. Σας αρκεί αυτή η διευκρίνηση. Μπορούμε να ψηφίσουμε τότε. Ποιος είναι υπέρ. Παρακαλώ ποιος είναι υπέρ. Λοιπόν, Δέκα υπέρ. Κατά παρακαλώ. Εννιά. Εγκρίνεται. Α, αποχές. Δεν ρώτησα ποιος απέχει. Δύο αποχές. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 67 Τσάιερ. Υπέρ παρακαλώ. Ζητώ συγγνώμη. Τα μπέρδεψα λιγάκι. Καταπίπτει 67. Λόγω της προηγούμενης τροπολογίας ψηφίσαμε. Θα πρέπει να ψηφίσουμε παρόλα αυτά την 17, την επόμενη τροπολογία. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί διάφορες τροπολογίες από την 17 μέχρι μέχρι την 35 προτείνω εγώ. Συμφωνείτε? Σωστά τα λέω. Υπέρ, υπέρ αυτών των τροπολογιών, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 36, άρθρο 87α νέο. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία του εισηγητή. Μπορείτε να μας την εξηγήσετε. Κάποιες πολιτικές ομάδες μου το υπέδειξαν. Δεν μας δεσμεύει όμως, παρόλο που παγώνει μια κατάσταση. Κανονικά ε, καλυπτόμαστε από μια νομοθετική πράξη, δεν χρειάζεται να το επισημαίνουμε και στον εσωτερικό κανονισμό. Ε, ψηφίζουμε υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα. Θα πρότεινα να ψηφίσουμε σε Λίδιν διάφορες τροπολογίες από την 37 μέχρι και την 51. Γιατί πρόκειται για κείμενα που ανήκαν στην έκθεση Κόρμπετ και είχαν εγκριθεί στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Συμφωνείτε? Υπέρ αυτών των τροπολογιών. κατά, αποχές, μία αποχή, εγκρίνονται. Άρθρο 124, παράγραφος 1 και 2 αλφανές προφορική τροπολογία, ο εισηγητής θα μας την παρουσιάσει. Αυτό είναι ένα σημείο που ανέφερε ο κύριος Φόξ στην αρχή της συνεδρίας όταν είπαμε ότι θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση και με την ΟΚΕ και με την Επιτροπή των Περιφερειών. Απλές τροπολογίες για να συμμορφωνόμαστε με τη συνθήκη και τις ε, γνωστές διαδικασίες. Υπέρ. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι. Βέβαια, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή η προφορική τροπολογία. Τώρα έχουμε μια νέα τροπολογία προφα... προφορική του εισηγητή, άρθρο 125, παράγραφος 1 και 2 αλφανές. Θα ήθελα να μας την παρουσιάσετε και αυτή την ε, προφορική τροπολογία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτή που ψηφίσαμε μόλις ήταν για την ΟΚΕ και αυτή είναι για την Επιτροπή των ε, Περιφερειών, το δύο πράγμα. Μπορούμε να ψηφίσουμε. ποιο είναι υπέρ. Παρακαλώ σηκώστε το χέρι όσοι είστε υπέρ. Κατά. Οχές. Εγκρίνεται. Τώρα, φτάσαμε στην τροπολογία 52. Υπέρ, παρακαλώ, υπέρ. Κατά. Δώδεκα Εγώ απέχω. Άλλος που απέχει. Τέσσερις αποχές. Πάμε στην τροπολογία 53. Άρθρο 132. Συγγνώμη ψηφίσαμε την 52. Τώρα πάμε στην 53. Τα αποτελέσματα δεν είπατε. Α, μα τα είπα. 12 υπέρ, 8 κατά και μία αποχή τελικά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Έχετε δίκιο, δεν τα, δεν τα είχα ανακοινώσει επίσημα τα αποτέλεσμα. Πάμε στην ψηφοφορία 53 άρθρο 132. Ποιος είναι υπέρ της 53. Κατά. Αποχές. Ομόφωνα εγκρίνεται. Α, όχι, με μία ψήφο κατά. Εγκρίνεται με μία ψήφο κατά. Πάμε στην τροπολογία τη συμβιβαστική για το άρθρο 132α το νέο όπου ο εισηγητής καλό θα ήταν μας πει κάτι. για τη συμβαστική τροπολογία 3. Πρόκειται για μια συμβαστική τροπολογία που αφορά τη συνεργασία μας με τις Εθνικές Βουλές. Υπάρχουν δύο λόγοι για την τροπολογία αυτή. Πιστε... Καταρχήν η αρχική πρόταση του κυρίου Μπρόκ, η αρχική τροπολογία ήταν υπερβολικά διεξοδική. Δεύτερον, θέλουμε κάποια ελαστικότητα στη διαπραγματεύση με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να μην προεξοφλούμε από τώρα τις ακριβεί λεπτομέρειες που θα διέπουν τη σχέση μας με τα εθνικά κοινοβούλια. Κάτι να λέμε στον εσωτερικό κανονισμό, αλλά όχι εξαντλητικά, όχι υπερβολικά διεξοδικά. Ναι, με να το περιλάβουμε στον εσωτερικό κανονισμό, αλλά όχι με την παραμικρή λεπτομέρεια, όπω προέβλεπε η αρχική τροπολογία Μπροκ. Κύριε ε, Πρόεδρε, αποδέχτηκα την προσπάθεια του εισηγητή να επιτύχει μια επικοδομητική προσέγγιση όσον αφορά την διακοινοβουλευτική συνεργασία όπως ορίζει και το πρωτόκολλο αλλά το πρόβλημα είναι πως εδώ πέρα εισάγεται η έννοια ενός δικτύου και δεν μου αρέσει αυτό. Η συνθήκη δεν λέει τίποτα για την μορφή που θα λάβει αυτή η συνεργασία. Και η έννοια του δικτύου ξαφνικά να εισάγεται εδώ μέσα στον κανονισμό νομίζω πως ε, δυστυχώς θα μας δεσμεύσει σε κάτι το οποίο τελικά μπορεί να αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε. Η συνθήκη λέει πως πρέπει να ε, γίνουν ε, συζητήσεις μεταξύ ημών και των εθνικών κοινοβουλίων για την κατάλληλη μορφή που θα λάβει αυτή η συνεργασία και πρέπει νομίζω να μείνουμε στη διατύπωση της ε, συνθήκης, των κανονισμό μας. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, καλύτερα να μην πούμε τίποτα σε αυτή την ε, φάση ε, για το ζήτημα αυτό. Όταν καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τα εθνικά κοινοβούλια, τότε μπορούμε να επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό στον κανονισμό. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πρόωρο. Ε, Κύριος Μέντες Τεβίγκο. Όντως είναι διαδικαστικό το θέμα. Θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι ο πρόεδρος Κλάους υπέγραψε τη συνθήκη. Ο κύριος Μπροκ θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως είναι μια σημαντική στιγμή Κάποιοι από μας έχουμε εργαστεί 10 χρόνια για αυτή την υπόθεση και πλέον είναι οριστική η συνθήκη και τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, οπότε είναι και ευτυχής η συγκυρία. Τώρα εδώ για τις ε, τροπολογίες μας. Δεν ξέρω, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, αν θέλουμε ένα τέτοιο δίκτυο. Με ένα τέτοιο δίκτυο είμαστε ένας από τους 28. Ένα κοινοβούλιο μεταξύ των 28. και αυτό στην έκθεσή μου ήθελα ρητά να το αποφύγουμε και να κάνουμε εμείς μια προσφορά, να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα καθοδηγούμε την ε, διαδικασία και μπορούμε να πούμε πως εδώ πέρα εντάξει δεν ξέρω αν είναι πολύ λεπτομερές η διατύπωση αλλά είναι η προσέγγιση τελείως διαφορετική και σας, σας ζητώ να το λάβετε υπόψη. Θεωρώ λοιπόν πως για αυτό τον λόγο πρέπει να βρούμε μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη Δεν ξέρω ποια θα είναι, αλλά θα επειδή τώρα το θέμα πρέπει να πάει στην Ολομέλεια, προτείνω εγώ στον εισηγητή να αποδεχτεί την ε, δική μου τροπολογία αλλά με, βάση τη δική μου τροπολογία να καταλήξουμε σε μια νέα διατύπωση για να έχουμε απλά μια διαφορετική αφετηρία. Γιατί ε, το Κοινοβούλιο είναι ένας από τους ε, δύο συνομοθέτες και όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν είναι ένας από τους 28, μην γίνει ένας από τους 28, ε, οπότε θα μπορούσαμε ίσως να δεχτούμε την κάπως ε, μακροσκελή δική μου τροπολογία, αλλά μπορούμε να κάτσουμε μαζί με τον ε, εισηγητή και να την σύντομεύσουμε λίγο, για να αλλάξουμε προσέγγιση δηλαδή. Ονορέουλε Μάρτιν. Κύριος Μάρτιν, Ντέβιτ είναι πρόταση αυτή. παρά είναι γενναιόδωρος ο Έλμαρ όπως πάντα. Εγώ θα πώς δεν θα υπερψηφίσω τις τροπολογίες με τη μορφή που έχουν. Εγώ νομίζω ότι υπήρχε συμφωνία για την συμβαστική λύση, αλλά φαίνεται πως όχι, γι' αυτό και την αποσύρω. Και ας αποφασίσει ο καθένας ε, πώς θα ψηφίσει στις τρεις τροπολογίες του Έλμαρ. Σε επίπεδο επιτροπή όμω ίσω τραβώσουν τα πράγματα. Θα μπορούσαν να δεχθούν μια προφορική τροπολογία στην 70 που λέει οποιαδήποτε έγγραφο που ε, επιδίδεται επίσημα από τα Εθνικά Κοινοβούλια στο Ευρωπαϊκό, να πούμε τουλάχιστον όποιο νομοθετικό έγγραφο ε, διαβιβάζεται επίσημα. Να προσθέσουμε και το νομοθετικό και να αφήσουμε το κάθε μέρος της Επιτροπής ε, εν τη σοφία του να λάβει θέση επί των τριών τροπολογιών του Έλμαρ. Αν κατάλαβα καλά, η τρίτη συμβιβαστική τροπολογία αποσύρεται. Έστω και προσωρινά. Και θα δούμε τι θα γίνει στην Ολομέλεια. Θα πρέπει να ψηφίσουμε την 68, 69 και 70. Και την 70 με τη διόρθωση που μας είπε ο εισηγητής. Σωστό? Μπορούμε να τις ψηφίσουμε και τις τρεις μαζί. Πολύ ωραία. Ποιος είναι υπέρ στις τροπολογίες 68, 69 και 70. Υψώστε τα χέρια. Κατά. Αποχή. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην υπερψήφιση των τελευταίων τροπολογιών από την 54 και μετά, μέχρι την 59 δηλαδή. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε σελίδι, νομίζω, αν δεν έχετε αντιρρήσει. Ποιο είναι υπέρ των τελευταίων τροπολογιών, κατά. Αποχές. Εγκρίνονται και τροπολογίες αυτές. Και τώρα θέλουμε να κάνουμε τελική ψηφοφορία για την πρόταση απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπέρ παρακαλώ. 19 υπέρ. Κατά. Δύο. Αποχές. Ένας. Απέχει. Εγκρίνεται. Και το έγγραφο συνολικά. Συγχαρητήρια κύριε Μάρτιν και εκ μέρου του Προέδρου θα ήθελα να συγχαρώ και τις Προεδρίας γενικά, θα ήθελα να συγχαρώ και τον κύριο Κόρπετ που προετοίμασε τις εργασίες. Νομίζω ότι τελειώσαμε την μέση διάταξη, έτσι δεν είναι. Τελειώσαμε, όντως. Για σήμερα το βράδυ θα τα πούμε αύριο το πρωί. Τώρα θα ξεκινήσει όμως η συνεδρία των συντονιστών. Ευχαριστώ.